με το θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Λάιτφριντ θα ξεκινήσει τέσσερα λεπτά ακριβώς, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε, στα τέσσερα λεπτά. Σε αυτό το νομοθετικό έργο πρέπει κανείς να πει περί τίνος δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε νέες προδιαγραφές όσον αφορά την μέτρηση της ηχητικής όχλησης ή του θορύβου στα αεροδρόμια. Δεν πρόκειται θέματα να εξετάζονται επιστημονικά διαφορετικά ή να αλλάξουν και να τροποποιηθούν. Όχι. Πρόκειται για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την πρόθεση να υπάρξουν κάποια μέτρα τα οποία με, σε ένα πιο ενιαίο πλαίσιο να μπορούν να εφαρμόζονται. Διότι είχε ανησυχίε σε διαφορετικά κράτη να υπάρχουν διαφορετικοί ε, γνώμονες και διαφορετική μέτρηση και κανόνες για την ηχητική όχληση. Θέλαμε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο και αυτό ήταν ο λόγος αυτής της προσπάθειας. Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί και συχνά όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπόψη κάτι, τότε πολλές φορές χάνει την αναγκαία αναλογικότητα και το σωστό μέτρο. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να διαρωτηθεί κανείς. Τι ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήθελε de facto ένα νομοθέτημα που θα δίνει τη δυνατότητα εθνικά μέτρα στα αεροδρόμια όταν δεν ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια να καταργούνται και υπήρξε μια διαμεσολάβηση πολιετής που ολοκληρώθηκε προς ικανοποίηση όλων. Η άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών ήταν ότι τέτοια μέτρα δεν θα είχαν νόημα. Ότι ακριβώς αυτό είναι το νόημα εκείνων που απορρίπτουν πολλοί πολίτες στην Ευρώπη. Δηλαδή ενοχλούνται πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε δεν πρέπει να εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ανακατεύεται σε θέματα που αφορούν εθνική νομοθεσία και εθνικές αρμοδιότητες. Στη συνέχεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο βρήκαμε μια λύση πιστεύω που καλύπτει αυτά τα θέματα και αυτές τις ανησυχίες και μελήματα και μεριμνά ώστε να μην υπάρχει μια δυσανάλογη ανάμειξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα εθνικών αρμοδιοτήτων και να μπορούν αυτά μελλοντικά να ρυθμίζονται έτσι, αλλά εκείνο το οποίο είναι δυνατόν να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει ενημέρωση και πληροφόρηση τι ακριβώς συμβαίνει και να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Είναι ένα πακέτο που έχει νόημα συνολικά και μπορεί να λειτουργήσει. Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν στόχος αυτού του νομοθετικού εγχειρήματος να ρυθμίσουμε τα πράγματα εκ νέου, να, τα, ε, ε, να νομοθετήσουμε διαφορετικά ή να δώσουμε διαφορετικές ερμηνείες. Άλλοι κανονισμοί και άλλες οδηγίες θα χρειαζόταν χρειαζόντουσαν για κάτι τέτοιο, αν κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο. Αλλά δεν ήταν έργο μας αυτό. Έργο μας ήταν να μεριμνήσουμε η αρχή της επικουρικότητας να διαφυλαχθεί και να ισχύει. Θέλω να δραθώ τις ευκαιρίες, μια και έχω τον λόγο, να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές. Ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η κοινή συνεργασία που είχαμε αναμεταξύ μας και καλό είναι αυτό. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα κοινού, κοινής προσπάθειας και κοινής εργασίας Καλό αυτό. Με σκληρή δουλειά κατα... μπορέσαμε να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν. It's... Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε Λάιχτφριντ. Ο Επίτροπος Κάλλας τώρα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Υποστηρίζω τη συμφωνία για τη μείωση τη ύπανση στα αεροδρόμια που επιτεύχθη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και σα παρουσίασε ο κύριος Λάιφτιτ. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον εισηγητή και τους και εισηγητές για τη σκληρή του δουλειά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καθοδηγήσει το τελικό αποτέλεσμα της μεγαλύτερης προβολής και των πτυχών της υγείας και το μεγάλο ε, βαθμό συμμετοχής ε, ε, του κοινού στην διαδικασία λήψης αποφάσεων λήφθηκαν αποφάσεις για αεροσκάφη τα οποία ε, συμμορφούνται προς, τους, ε, προς τις προδιαγραφές ε, οριακά και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν και περιορισμοί του θορύβου και κατάλληλα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι οι νέοι κανόνες ε, για τη ε, μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια αποτελούν καλό συμβιβασμό και θα προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες κατά της ηχητικής ρήπανσης, τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες θα αποφασίσουν τελικά για τα μέτρα τα οποία θα επιβληθούν σε κάθε αεροδρόμιο. Οι κανόνες ε, για το θόρυβο θα πρέπει ε, να βασίζονται στις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη ώστε ε, να συμμετέχουν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να λαμβάνονται αποφάσεις βάσει στοιχείων και βάσει του κόστους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές πρακτικές συμμορφούνται με τις αρχικές πρακτικές του ΑΙΚΑΟ, δηλαδή της ισορροπημένης προσέγγισης όπως αποκαλείται και θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και την ε, ε, Συμφωνία Μεταφορών Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών καταλήλως. Ε, αναφέρθηκε επίσης και η αναθεώρηση της οδηγίας για τον ε, περιβαλλοντικό θόρυβο και η δήλωση αυτή επισημαίνει πόσο σημαντική είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υγεία όπως ε, ε, γνωρίζω ότι είναι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Προεδρεύων, ευχαριστούμε Επίτροπε Κάλλας. Ακολουθούν τώρα οι αγορητές εξονομάτων των ομάδων. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος Γκάλερ παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η συμφωνία για τους κανόνες και διατάξεις ε, όσον αφορά τις ρυθμίσεις σε αεροδρόμια είναι μια, ε, μια καλή είδηση για τους πολίτες της Ευρώπης ιδιαίτερα για όλους εκείνους τους περιοίκους που κατοικούν σε μια περιοχή όπου λειτουργεί ένα αεροδρόμιο για παράδειγμα όπως ε, για μένα στη Φραγκφούρτη το αποφασιστικό στοιχείο το οποίο τονίστηκε από τον εισηγητή είναι ότι η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει πλήρως να μπορέσει να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί και με την ισορροπημένη προσέγγιση balanced approach να μπορέσει να λειτουργήσει. Εκεί όπου υπάρχει θόρυβος που προκαλείται και πρέπει να καταπολεμηθεί, οι αρμόδιες αρχές να έχουν το τελευταίο λόγο καλά ή θετικά επιχειρήματα ή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής σίγουρα ευχαρίστω θα τα λάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόψη. όμω η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται επιτόπου από τι αρμόδιε αρχέ. Και είναι σημαντικό και ήδη προαναφέρθηκε η προστασία τη υγεία να κατοχυρώνεται από πλευρά κειμένου και μια επεξήγηση δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει για τον κίνδυνο τη ηχητική όχληση στην υγεία, για τον θόρυβο περιγύρου που πρέπει και να λαμβάνεται υπόψη. Είναι καλή είδηση και αυτή για τους περίοικους, για εκείνους που κατοικούν κοντά σε αεροδρόμια, που τα ιδιαίτερα ηχητικά, οχλητικά αεροπλάνα να μπορούν να περιορίσουν το θόρυβο αυτό και να μεριμνήσουμε οι περίοικοι να μπορούν στο μέλλον να προστατεύονται και να ενημερώνονται ακόμα καλύτερα για ό,τι σχεδιάζουν από πλευράς αεροδρομίων και αεροπλάνων και κίνησης αεροπλάνων. Είναι καλό αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να μεριμνήσουμε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους αρμόδιους επιτόπου να διασφαλίζεται και η διαδικασία διαμεσολάβησης που σε πολλούς τομείς είναι σημαντική να κρατήσει αυτή την αξία της. Ευχαριστώ όλους που συνεργάστηκαν σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Προεδρεύων, ευχαριστούμε συνάδελφε Γκάλερ. Για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Λιντεράτσκι παρακαλώ. Μικρόφωνο. Με μικρόφωνο παρακαλώ κύριε Λιντεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί έχει ετοιμάσει εξαίρετο εγγραφό. Συγχαρητήρια λοιπόν για την επιτυχία αυτή εδώ, όταν ο κύριος Κάλας προσωπικά συμφώνησε πως τα επιχειρήματα που προωθούνται είναι σωστά. Περισσότερη ευελιξία για τις χώρες μέλη, περισσότερη μέρημνα για τα θέματα υγείας και περισσότερη ανάμιξη όσων ζουν κοντά σε αεροδρόμια. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά η επιτυχία είναι διασφαλισμένη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να είναι αποφασιστική σημασίας και ο κύριος Σκάλας συμφώνησε με τα επιχειρήματα αυτά. Όχι πάρα πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αρκετή Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα που είναι σημαντικά. Είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και πολλοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει το ένα, μας επιβάλλει το άλλο. Ναι, αλλά μερικές φορές λύνει προβλήματα. Πάντως η πρωτοβουλία πρέπει να είναι στα χέρια των πολιτών μας. Ήδη λοιπόν έχουμε μια επιτυχία για αυτό το θέμα. Τέτοια θέματα πρέπει να αναφέρονται τα επίπεδα ζωής, οι συνθήκες ζωής και χαίρομαι που αναφέρονται εδώ. Όμως δεν ρυθμίζουμε τα μικρά αεροδρόμια και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι στέκει. Προεδρεύω, σας ευχαριστούμε, συνάδελφε Λιβεράτσκι. Συνάδελφος Μάισνερ, 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή ε, τον κύριο Λάιχφριντ. Ο συνάδελφος ο οποίος θέλει να εκφράσει ευχαριστίες του σήμερα δεν μπορεί να παραστεί και τις εκφράζω εγώ εξ ονοματός του. Πολλά αναφέρθηκαν. Φυσικά είναι το ότι χρειαζόμαστε τις εναέριες μεταφορές. Οι εναέριες μεταφορές είναι πολύ σημαντικές για την Ευρώπη και πολλοί λένε θα αυξηθούν κιόλα. Πρέπει να σκεφτούμε να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των μεταφορών και να δημιουργηθούν τέτοιε προϋποθέσεις για τα αεροδρόμια εκείνοι που κατοικούν κοντά στα αεροδρόμια να μην ε, ε, υφίστανται την ηχητική όχληση ε, σε διαστάσεις που δεν είναι πλέον ανεκτές. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε επιτόπου πώς μπορεί να διασφαλιστεί όλα να γίνουν για να προστατευτεί η υγεία των περίοικων αλλά και να υπάρξει το πλαίσιο για τις μεταφορές που θα διασφαλίσει και τις θέσεις απασχόλησης όπως χρειαζόμαστε. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι αναγκαίο. Και για παράδειγμα σήμερα μιλήσαμε για εναλλακτικές πηγές ενέργειας να σκεφτούμε το αεροδρόμιο του μέλλοντος θα μπορούσε ίσως την κινητικότητα, την ηλεκτρική κινητικότητα να την εκμεταλλεύεται σε αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό θα περιόριζε την ηχητική όχληση. Είναι όμως θέματα που αφορούν το μέλλον αυτά και όχι σήμερα το παρόν. Θα πρέπει όμως επιτόπου να μπορούν να αποφασιστούν αυτά τα θέματα και να λύνονται τα προβλήματα. Όχι στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις επιτόπου και επιτόπου πρέπει από τους πολίτες να μπορούν να λύνονται τα προβλήματα και να λαμβάνονται οι αποφάσει. Ευχαριστώ. Προεδρεύον, ευχαριστούμε συνάδελφε Μάισνερ. Λίχτενμπεργκερ, ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κυρίω τον συνάδελφο Λάιχτφρεντ που από κοινού με όλους εμάς σε ιδιαίτερο βάθος διαπραγματεύτηκε και συζήτησε. Και ευχαριστώ σε αυτή την περίπτωση και το Συμβούλιο που ενέκρινε, έδωσε την έγκρισή του. Και καταφέραμε να έχουμε, <clears throat> για παράδειγμα, να αποφύγουμε μία παρέμβαση στις αρμοδιότητες των τοπικών αρχών στα θέματα αεροδρομίων. Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Όποιοι το γνωρίζουν, το αξιολογούν σωστά. Χρειάζεται και εδώ υιοθετείται δυστυχώς η ε, balanced approach, η ισορροπημένη προσέγγιση γιατί λέω δυστυχώ, διότι balanced approach θα σημαίνει δεν θα υπάρχει περίοδος νυχτερινή ησυχία, αλλά θα υπάρχουν κάποια παράθυρα προστασίας από την ηχητική όχληση. Δηλαδή κάποιες μικρές χρονικές περίοδοι προστασίας από την ηχητική όχληση των αεροπλάνων που προσγειώνονται και απογειώνονται. Όταν αρχίζουμε να σταθμίζουμε τέτοιου είδους πράγματα, τα συμφέροντα δηλαδή των επιχειρήσεων, πορευόμαστε είμαστε σε σφαλμένη τροχιά. Όλα μπορεί να είναι σημαντικά τα θέματα των βιομηχανιών, των επιχειρήσεων, αλλά έχω τεράστιες επιφυλάξεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Στη συνέχεια η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συμμορφόμαστε ήδη στην ισορροπημένη ε, απόφαση του ΙΚΑΟ και έχει μειωθεί ο θόρυβος. Προσπαθούμε επίσης να επιταχύνουμε τους ενιαίους ευρωπαϊκούς θέρες. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τους κινητήρες. Πρέπει να τα ενθαρρύνουμε όλα αυτά, να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε βέβαια κάποιες ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούσε η έκθεση αυτή και τώρα χαίρομαι που μπορώ να πω ότι αντιμετωπίστηκαν οι ανησυχίες μας αυτές γιατί η επικράτησε κοινή λογική και τηρήθηκε η επικουρικότητα. Συνεπώς, η πρόοδος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν πολύ σημαντική, οπότε η ομάδα μου, το ECR, θα μπορέσει με χαρά να στηρίξει τη ρύθμιση αυτή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους και τους σκιώδεις εισηγητές που συνεισέφεραν σε αυτό. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ πολύ κύριε Λάχτφριντ. Πρόεδρος, κυρία Φώστα, συνάδελφε Φώστερ, επιτρέπετε μια επερώτηση του κυρίου Ρούμπιχ. Μια μπλε κάρτα του κυρίου Ρούμπιχ. Κύριε Ρούμπιχ, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά Πρόεδρε γι' αυτό. Η ερώτησή μου αφορά τις προσπάθειες έρευνας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Horizon 2020, ορίζοντα 2020 και τις δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν και θέματα εναέριων μεταφορών. νομίζετε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, έχετε τον λόγο να απαντήσετε. Ναι, το κυριότερο είναι ότι έχουμε το Clean Sky που είναι μια κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία που προσφέρει πολλά για την επόμενη γενιά αεροσκαφών με πολλά εκατομμύρια επενδύσεις. Πιστεύω ότι θα επιταχυνθεί η εφαρμογή και του ΣΕΖΑΡ και των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων. Αυτός είναι ο δρόμος μπροστά. Έχουμε τα μέσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φώστερ. Δεν υπαρίσταται ο κύριος Κόχλιτσεκ. Ο κύριος Μαρινέσκου παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αηφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών επιβάλλει να, βάλουμε, να λάβουμε υπόψη μας διάφορα μέτρα για να μειώσουμε την ηχορύπανση στα αεροδρόμια. Με τη ρύθμιση του ΙΚΑΟ έχουμε οδηγηθεί σε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Η αρχή είναι, που περιλαμβάνεται και στη Συμφωνία του Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου, να μειωθεί ο θόρυβος των αεροσκαφών, αλλά να υιοθετηθούν και μέτρα για καλύτερη διαχείριση του χώρου γύρω από τα αεροδρόμια, ώστε να υπάρξουν και μειώσεις λειτουργικού χαρακτήρα. Τα μέτρα που προτείνονται είναι ισορροπημένα και τηρείται και αρχή της επικουρικότητας. Δεν πρόκειται για ριζοσπαστικά μέτρα, δεν θα καταστραφεί η αεροβιομηχανία δεν επιβάλλει μείωση της κυκλοφορίας παρά μόνο εφόσον ο θόρυβός τους βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Είναι μια αρχή πρόληψης. Και δίνει και όθηση για εξυγχρονισμό στην βιομηχανία στους κατασκευαστές αεροσκαφών. Πάντως οι χώρες και οι περιφέρειες μπορούν να συναποφασίζουν γιατί είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τους ίδιους κανόνες παντού σε όλα τα αεροδρόμια που διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους ανάλογα με το που βρίσκονται και πώς είναι φτιαγμένα και τι μεγέθους είναι. Μην ξεχνάμε ότι θέλουμε και την ανάπτυξη των περιφερειών όπου βρίσκονται τα αεροδρόμια. Ο ρόλος τους είναι δύσκολος γιατί πρέπει να δουν συνολικά το θέμα η αεροναυπηγική είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ασφαλή απασχόληση αν δεν επιτρέψουμε στον τομέα να διασφαλίσει προστασία για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Μαρινέσκου. Περνάμε στη διαδικασία κάτω στη παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Eh, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Οι περιορισμοί για το θόρυβο στα αεροδρόμια είναι ένα πάρα πολύ καλό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε διαμακρών και μπορέσαμε, ε, σύντομα θα το εγκρίνουμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται όλους τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες οι οποίοι επιβαρύνονται από τα αυξημένα επίπεδα θορύβου και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και περιορισμοί στις νεκτερινές πτήσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Συμβούλιο να μην προσπαθήσει να ενερμανίσει τα πάντα. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονό ότι δεν προσπαθεί να ενερμανίσει τα πάντα. Ε, πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή τη επικουρικότητα και θεωρούμε ότι θα πρέπει όμω ταυτόχρονα να λαμβάνουμε υπόψη και του κινδύνου για την υγεία των πολιτών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία με την κυρία Τίκαου. Ε, subliniez importanța επισημαίνω την ε, μεγάλη σημασία της εναρμόνισης και της διευκρίνησης των κοινών κανόνων όσον αφορά τους περιορισμούς ε, για τον περιορισμό των ηχητικών οχλήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Χαίρομαι που οι τοπικές αρχές θα έχουν και το δικαίωμα απόφασης για το ποσοστό της μείωσης των θορύβων και τα σχετικά μέτρα και μέτρα για τις νεκτερινές πτήσεις. Ε, όσον αφορά τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θορύβων, υποστηρίζω την αναθεώρηση τη σχετική οδηγία και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα προσέξει συγκεκριμένε λύσει για τα προβλήματα υγεία που προκαλούνται από την ηχορύπανση στα αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Τίκα. Ο επίτροπο Κάλλα, παρακαλώ έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας η συζήτηση αυτή καταδεικνύει ότι όντως μπορούμε να επιτύχουμε ε, καλά αποτελέσματα για τους ελέγχους στα αεροδρόμια. Η έγκριση του κανονισμού για τη μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια θα ανοίξει και το δρόμο για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του νέου ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα σλότς των αεροδρομίων και άλλα θέματα που αφορούν ε, τη δέσμη μέτρων για τα αεροδρόμια. Ο κανονισμός για το θόρυβο αποδεικνύει ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όσον αφορά την έρευνα, κυρία ε, Φώστερ, που αναφέρατε, συνεισφέρουμε σημαντικά στον ενίο ουρανό, στο Single Sky, σε ό,τι έχει σχέση με τον ενίο ουρανό, ε, συνεισφέρει άλλωστε και στη μείωση της ρήπανσης και της συγχωρήπανσης. Και ε, σίγουρα θα συνεισφέρουμε και στην έρευνα και στην ανάπτυξη για κινητήρες οι οποίοι θα βοηθήσουν ε, τη μείωση των θορύβων και χαιρόμαστε που η έρευνα σε θέματα μεταφορών θα χρηματοδοτείται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ε, στις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε Κάλλας. Ολοκληρώνεται η διαδικασία με την παρέμβαση του συναδέλφου Λάιχτφριντ. Τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ότι τη ουσία σχεδόν όλα αναφέρθηκαν. Θέλω να δραχθώ και πάλι τις ευκαιρίες και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που επικοδομητικά συνεργάστηκαν για αυτή την νομοθετική πρόταση. Θέλω επίσης και πιθανότατα είναι ο τελευταίος μου κοινοβουλευτικό λόγος που εκφωνώ σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να μου επιτρέψετε μια παρατήρηση. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ, συνάδελφοι, που είναι πάντα εναντίον όλων. Ποτέ δεν εργάζονται και δεν συνεργάζονται σε κάποιες προτάσεις. Το κύριο έργο τους είναι, εδώ στην Ολομέλεια, να διαμαρτύρονται. Είναι υπέρ του περιορισμού των δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου και μάλιστα και υπέρ της κατάργησης του Ευρωκοινοβουλίου. Αν τώρα δει τα αποτελέσματα κανείς που έχουμε εδώ ενώπιόν μας σε σχέση με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε καλύτερο νομοθετικό έργο το οποίο προκάναμε σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπεύθυνοι για το ότι δεν μπορούν οι πολίτες της Ευρώπης να καθορίζουν ποιοι αποφασίζουν για την συνυπευθυνότητα στο νομοθετικό έργο. Είναι κατά της δημοκρατίας στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι και εγώ είμαι κατά αυτών. Είμαι υπέρ ενός ισχυρού με συνειδητοποίηση κοινοβουλίου που θα μεριμνά για περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη και θα την δημιουργεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε συνάδελφε Λάιφρυντ. Ολοκληρώθηκε έτσι η συζήτηση εδώ. Η έγκριση, η ψήφιση θα γίνει κατά την ψήφιση την Τετάρτη και το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση για τα τρόφιμα και τα, τις ζωοτροφές και την υγεία των φυτών. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Πυρίλο. Νομοθεσία για τα τρόφιμα, της ζωοτροφές, κανόνες για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, υγεία φυτών, την έκθεση της κυρίας Πάουλσεν. υγεία των ζώων και